την Επιτροπή αυτά δεν τα θεωρούμε απλώς καθήκον ή υποχρέωσή μας. Με μεγάλη χαρά ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για το θέμα της απόψινής συζήτησης. Ε, ο, έκλεισε εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή με θέμα ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της κοινότητας. Ε, ξεκινούμε τη συζήτηση. Το λόγο θα πάρουν οι συντάκτες της ε, ερώτησης. Ο κύριος Λίζη έχει πρώτος το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Το 2008 είχαμε σημαντικές ε, διαπραγματεύσεις για την ενσωμάτωση των αεροπορικών μεταφορών στο σύστημα ανταλλαγής εκπομπών αερίων. Εγώ ήμουν συντάκτης ε, της έκθεσης και πολλοί από τους ε, συναδέλφους που συνέπραξαν σε αυτήν εδώ παρόντες. Το σύστημα λοιπόν αυτό το εισαγαγαμε όχι γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα είτε στην αεροβιομηχανία είτε στις ξένες αεροπορικές εταιρείες αλλά γιατί έχουμε να κάνουμε ένα πραγματικό πρόβλημα. Ξέρουμε ότι έχουν διπλασιαστεί μέσα σε πολύ λίγα χρόνια οι εκπομπές ε, των αερίων θερμοκηπίου. Το 1997 λοιπόν προσδιορίστηκε ο, ε, η ανάληψη των αρμοδιοτήτων από την ε, ΙΚΑΟ για προσδορισμό των συνθήκων περιορισμού των εκπομπών ε, καυσερίων από τα ε, αεροπλάνα, πράγμα το οποίο όμως ακόμα δεν έχει γίνει. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με, αεροπλάνο, με ένα σύστημα το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε είδους αεροπλάνο που προσγειώνεται ή απογειώνεται σε ή από ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, είτε πρόκειται για εταιρεία ευρωπαϊκή, αμερικανική, κινέζικη ή άλλη. Το, σύστημα δηλαδή, το, το, το, το ζήτημα είναι δηλαδή το σύστημα να εφαρμόσει σωστά. Έχουμε κάνει πολλές, ε, πολλούς συμβασμούς μέχρι τώρα. Πρέπει όμως πλέον να εξηγήσουμε και στα τρίτα κράτη ότι δεν μπορούν αυτοί οι συμβασμοί να ε, συνεχίζονται επαόριστον. Βρισκόμαστε σε δικασία συναπόφασης. Είχαμε μέχρι τώρα ε, την εξαγγελία από τρίτα κράτη ότι πρόκειται να προσφύγουν στην ΕΚΑΟ, τη οποία η Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει την προσεχή εβδομάδα. Εγώ θεωρώ και έχω μελετήσει πολύ το θέμα ότι νομικά είμαστε καλυμμένοι. Το θέμα όμω πάνω απ' όλα είναι πολιτικό. Και γι' αυτό χρειάζεται και πολιτική κάλυψη από του και για του διαπραγματευτέ μα, εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Επίτροπο Κάλλα και εκ μέρου βέβαια του Συμβουλίου, την ε, Βελγική Προεδρία. Ε, οι Αμερικανοί, παραδείγματι, ξέρουμε ότι θα πιέσουν ιδιαίτερα. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα να συναντήσω τον αρχιδραματευτή των Αμερικανών και τον ρώτησα εάν θεωρεί ότι μπορεί να ε, συνάδει η στάση τους στην ΙΚΑΟ με τα όσα έχει αποφασίσει και το Κογκρέσο αλλά και τα όσα έχει δηλώσει και εξαγγείλει ο πρόεδρος Ομπάμα γιατί εάν ε, ε, δράσουν κατά αυτόν τον τρόπο που ε, εξαγγέλουν θα πρέπει ουσιαστικά να αναιρέσουν τα όσα έχει αποφασίσει το Κόγκρεσο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκρότε Ματίας για τρία λεπτά. Μην ξεπεράσετε το χρόνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Στην 11 ώρα ήρθαμε να συζητήσουμε το κλίμα μέσα σε συνθήκες οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουμε πολλά προβλήματα φυσικά αλλά και οι κλιματικές αλλαγές ε, και την προστασία του κλίματος έχει τεράστια σημασία και νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί ενδιαφέρονται να μάθουν πώς θα χειριστεί το ζήτημα στην πραγματεύση της ΕΚΑΟ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπε και ο κύριος Λύση έχουμε αγωνιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στο Κοινοβούλιο έτσι ώστε οι αεροπορικές μεταφορές να ενταχθούν στο σύστημα της ανταλλαγής εκπομπών ε, ε, καυσαερίων. Έχουμε πολλές φορές διαπραγματεύεται τα θέματα αυτά και με το Συμβούλιο και πρέπει αυτά που έχουμε αποφασίσει να τα προβάλλουμε και προς τα έξω και να τα υποστηρίξουμε και στις ε, διεθνείς μας ε, επαφές και διαπραγματεύσεις. Για τον περιορισμό λοιπόν των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα έχουμε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, τα αποτελέσματα όμως σε επίπεδο ΙΚΑΟ είναι μηδενικά και γι' αυτό πιστεύω ότι η δική μας πρόταση, αυτή την οποία με τόσο ευρία πλειοψηφία υιοθετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει πιστεύουμε να ισχύσει και να προαχθεί σε διεθνές επίπεδο. Από το 2012 και μετά αρχίζει να ισχύει το, το σύστημα αυτό στο οποίο θα εντάσσονται και τα τρίτα τα αεροπλάνα από τρίτα κράτη ε, είτε προσγειώνονται είτε απογειώνονται ε, σε ή από ευρωπαϊκό αεροδρόμιο θα πρέπει να εντάσσονται σε αυτό το σύστημα. Το κλίμα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και έτσι πρέπει να είναι παγκόσμιες και οι λύσεις που θα δοθούν. Εάν κανείς διαφωνεί και δεν θέλει να υπαχθεί σε αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κάποια συστήματα ε, με τέλη ή με οικονομική πίεση τα οποία, ή με φόρο ενδεχομένω τα οποία θα ε, μπορούν να ε, πιέσουν προς την κατεύθυνση αυτή. Εάν επιβληθεί ρηβγόνος φυσικά θα υπάρχει καμιά εμβολία ότι πρόκειται για φόρο για το δεξίδιο του άνθρακα. Πιστεύουμε ότι η, καλύτερη, η δεύτερη, αν θέλετε, καλύτερη λύση είναι αυτή της ένταξη των ε, αεροπλάνων τρίτων κρατών στο σύστημα της ανταλλαγής των ε, καυσαερίων, το οποίο ελπίζουμε ότι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, το οποίο λάμπει τέτοια ώρα δια τη απουσία του, να υποστηρίξει και στι διεθνεί διαπραγματεύσει. Διεθνεί φορεί και παράγοντε είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η κυβέρνηση Ομπάμα ξεκίνησε με πολύ μεγάλου και υψηλού στόχου όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ. Στόχου όμω που πέραν των διακηρύξεων δεν είδαμε να εφαρμόζει στην πράξη. Και εδώ βλέπουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε νομοθεσία για το κλίμα που να τη φέρει σε επίπεδο ισοδύναμο με το δικό μας ή σε υψηλό επίπεδο παγκοσμίω. Κινδυνεύουμε λοιπόν, εάν δεν συμπράξουν οι Αμερικανοί, το ζήτημα αυτό να πέσει στο νερό. στο σύστημα της ε, ικαο στη συμφωνία της ικαο υπάρχει ολόκληρη η συμφωνία για τις κλιματικές αλλαγές και θα ήθελα να ρωτήσω την ευρωπαϊκή επιτροπή εάν δεν υπάρξει συμφωνία ως προς τις, ε, κλιματικές, εκπομπές μέσα και την υπαγωγή ε, των αεροπορικών μεταφορών σε αυτές. Υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουν μια διέξοδο και ένα διαφορετικό σχέδιο εάν αυτά αποτύχουν. παρακαλώ πολύ να είστε πολύ προσεκτικοί στα περιθώρια που έχουμε γιατί πρέπει να τελειώσουμε στην ώρα μας. Ο κύριος Κράμερ για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δυστυχώς σήμερα έχουμε να συστήσουμε μια αποτυχημένη στρατηγική. Ήταν αποτυχημένη από τη στιγμή ήδη που υιοθετήθηκε η οδηγία. Ήδη την ώρα που τη συζητούσαμε βλέπαμε πότε θα εκπνεύσει γιατί δεν εντάσσονται στο σύστημα της ανταλλαγής των εκπομπών τα τρίτα κράτη. Και φαίνεται ότι και σήμερα ακόμη αγνοούμε την κατάσταση όπως ισχύει διεθνώς. Βλέπουμε ότι και η συνέχεια της Κοπεχάγης ε, με τη διάσκεψη ΚΑΟ δεν πρόκειται να προχωρήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να δούμε τη λύση μιας ευρωπαϊκής οδηγίας που πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκοπεύει να κάνει. Περιμένω με αγωνία να ακούσω την απάντηση ποια είναι τα μέτρα τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επιβάλλει σε ε, αεροπορικές εταιρείες ή σε, αεροπλ... κράτη τρίτα, τα οποία δεν υπάρχονται στο σύστημα αυτό. Πώς μπορεί να επιβάλλει το σύστημα των ανταλλαγών. Πώς μπορεί να ε, επαληθεύσει ή να σχεδιάσει ε, μέτρα για τις ε, αεροπορικές εκείνες εταιρείε στα τρίτα κράτη τα οποία αρνούνται να επαχθούν στο σύστημα των ανταλλαγών και σε περίπτωση που, επιβληθούν ε, απαγορεύσεις ε, πτήσεως τι αντιδράσει περιμένει η Επιτροπή από τα τρίτα κράτη. Σημειώνω ότι υπάρχουν και σχετικέ δικαστικέ υποθέσει από κράτη και αεροπορικέ εταιρείε, οι οποίε αντιδρούν και δεν δέχονται να υπαχθούν στο σύστημα αυτό. Τι θα γίνει λοιπόν από το 2012 και μετά. Το πώς θα χειριστούμε τις διαπραγματεύσεις μέσα στην ΙΚΑΟ για μένα είναι λίγο πολύ δευτερεύουσα σημασίας. Γιατί πρέπει να περιμένουμε ε, λίγο πολύ αντίστοιχε αντιδράσει με αυτέ που είδαμε στην Κοπενχάγη από τα τρίτα κράτη. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ εγώ την Επιτροπή το δίλημα αυτό Πώς θα το ξεπεράσουμε, πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να εφαρμόσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο ουσιαστικά δεν είναι εφαρμοστέο, δεν είναι εφαρμόσιμο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Hyvät kollegat, lentoliikenteen päästöt ovat kasvaneet έχει αυξηθεί η εμπορία ε, εκπομπών σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Διπλασιάστηκαν σε 20 χρόνια. Η... Εάν, παρόλο που γίνονται προσπάθειες να μειωθούν τα, οι εκπομπές αυξάνονται στον τομέα της, ε, των αεροπορικών μεταφορών το, η συμφωνία του Κιώτο υπεγράφει ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών. Αλλά δεν πέτυχε το στόχο της αυτή η συμφωνία. Θέλουμε να ε, ισχύσει ένα παγκόσμιο σύστημα. Αλλά το σύστημα εμπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπωσδήποτε έχει ευρύτερη, ευρύτερη επιρροή. Τα αεροσκάφη που φτάνουν στην Ευρώπη αποτελούν σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας πολιτικής αεροπορίας. Πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πίεση Οπωσδήποτε αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα που έχει ο πρόεδρος Ομπάμα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από το Κογκρέσο της χώρας του για να περάσει ορισμένα ε, νομοθετήματα για να σώσει τον πλανήτη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε ωστόσο στις Ηνωμένε Πολιτείες να, ακολουθεί, να εξακολουθήσει να ακολουθεί μια τέτοια πολιτική πρέπει, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε Κάτι αντίστοιχο άλλωστε ισχύει και την ε, διεθνή ναυτιλία. Πρέπει να τηρήσουμε τις αποφάσεις που έχουμε λάβει. κύριος Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα εκ μέρου του συναδέλφου Κλοντ Χέντικατ που ασφαλώς θεωρεί πολύ σημαντικό ε, το ζήτημα αυτό και έφθετο το χρονικό σημείο στο οποίο υποβάλλεται η ερώτηση. Δυστυχώ δεν μπόρεσε να έρθει γιατί βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τι συναντήσει των ΗΠΑ. Ε, έχουμε λοιπόν τη σύνοδο από τις 28 ε, Σεπτεμβρίου, ξεκινάει 28 Σεπτεμβρίου, με το θέμα αυτό το οποίο συζητούμε την ε, προηγούμενη εβδομάδα το Συμβούλιο της ΚΑΟ ε, προσπάθησε να ε, περάσει ένα σχετικό ψήφισμα αλλά δεν τα κατάφερε. Ο μονομερής στόχος του περιορισμού του οξυδίου του άνθρακα στο 20% κάτω από το επίπεδο του 1990 είναι ένα στόχος τον οποίο ακόμη δεν, δεν αντικαθιστά κανένας άλλος διεθνής στόχος και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει έτσι. Οι εκπομπές φαίνεται ότι θα εξακολουθήσουν να αυξάνονται και θα είναι κατά 70% ε, υψηλότερες από ότι το 2005 όπου μιλούσαμε για ανταλλαγές 4 με 5% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ιδιαίτερη σημασίας απόφαση που το 2008 από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, με την εισαγωγή των αεροπορικών εταιριών που προβλέπεται από το 2012. Αυτό ισχύει, 12. Αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις αεροπορικές ε, εντός αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ξεκινήσει η προεργασία, θα πρέπει δηλαδή να συμβάλλουν όλες τις εταιρείες στο σύστημα για την προστασία του κλίματος με ε, ισοδύναμα, ή αλλιώς με ισοδύναμα συστήματα τα οποία βοηθούν στον περιορισμό των εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο στις διαπραγματεύσεις επίπεδο ΙΚΑΟ μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις θέσεις μας τον ε, στόχο για περιορισμό των εκπομπών από τις αεροπορικές μεταφορές κατά 10% στο 2020 ε, μέτρα προσαρμοσμένα συνθήκες αγοράς για τον περιορισμό των εκπομπών μέσα από την ΕΚΑΟ και είναι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση διατεθειμένη να αποκλείσει από την εφαρμογή των μέτρων των ευρωπαϊκών ε, χώρα, τρίτη χώρα, η οποία εφαρμόζει ένα ισοδύναμο σύστημα. Ξέρετε όμως ότι διαφωνούν κυρίες και κύριοι οι ΗΠΑ και άλλα μέλη της ΕΚΑΟ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, προβάλλουν ε, ως λύση την ιδέα της αμοιβαίας συμφωνίας ε, η οποία όμως η οποία σε στόχο έχει μόνο να καταρρύψει το ευρωπαϊκό σύστημα. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε βέβαια να υπονομευθούν τα ευρωπαϊκά μέτρα από τους εταίρους μας στην ΕΚΑΟ γιατί πιστεύουμε ότι συμβάλλουν ιδιαίτερα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Δεν μπορούμε να δεχθούμε εκείνοι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν περισσότερο ή να, αγωνιστούν περισσότερο για τις κλιματικές αλλαγές να αντιμετωπίσουν προβλήματα από εκείνους που δεν θέλουν να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε αποτελεσματικά μέτρα για την κλιματική αλλαγή τα οποία μετατρέπονται σε μειονέκτημα ανταγωνιστικό για τις ε, χώρες μας και ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι αν εφαρμόζαν τα μέτρα αυτά χωρίς ένταξη και των τρίτων ε, κρατών και των, των, των εταιριών τους θα ε, βρίσκονταν οι ευρωπαϊκές εταιρείε σε ε, μειονεκτική θέση ανταγωνιστικά. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και οφείλει ουσιαστικά να προχωρήσει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και δεν είναι δυνατόν ευρωπαϊκή νομοθεσία μα από το, που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να ανατρέπεται από τρίτες χώρες ή παράγοντες. Στόχος μας είναι ο περιορισμός των εκπομπών, η, βράχη, η μέσοπρόθεσμη και διαρκής ε, περιορισμός των εκπομπων η η η μεσοπροθεσμη και διαρκης περιορισμος των καυσέριων. Των πολιτικών ομάδων. Για την ε, ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ο κύριος Ελκαντράουι για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την σαφέστατη απάντησή σας και για τις σαφείς απόψεις σας. Πιστεύω ότι ως Κοινοβούλιο πρέπει να στείλουμε, να απευθύνουμε ένα σαφέστατο μήνυμα, ένα μήνυμα υποστήριξης στην Επιτροπή. Διότι αν πιστεύουμε ότι η οδηγία ε, ε, ήρθε πολύ νωρίς ή πολύ αργά ή δεν προχωράει αρκετά, έχουμε πλέον θεσπίσει κάτι το οποίο αποτελεί νομοθεσία και πρέπει να εφαρμοστεί και εσείς πρέπει να αναλάβετε την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας ως Επιτροπή. Αυτή η νομοθεσία είναι σαφής, αναφερθήκαμε σε αυτή και λέει ότι από την 1η ε, Ιανουαρίου του 2010 για όλες τις πτήσεις που φεύγουν ή φτάνουν σε αεροδρόμιο ε, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία και συμπεριλαμβάνονται τα αεροσκάφη που έρχονται από τρίτες χώρες για την πτήση προς και από. Είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι γεγονός ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες εκφράζουν, διατυπώνουν κάποιες αμφιβολίες. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην ισχύει αυτό για τις τρίτες χώρες μόνο για τη μισή πτήση την ε, ε, ε, άφηξη ή επιστροφής ότι αυτό θα δημιουργούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού ανάμεσα στι αεροπορικές εταιρείε. Όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι οι αεροπορικές εταιρείε δεν είναι δυνατόν να μην υποβληθούν σε αυτά τα μέτρα και οι χώρες αυτές πρέπει να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Εάν όλοι ακολουθούσαν το παράδειγμά μας θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. Και αυτός άλλωστε είναι ο σκοπός αυτής της νομοθεσίας και οι Αμερικανοί φίλοι μας, ή άλλοι που επικαλούνται κάποιες ε, άλλες διατάξεις ή ε, χρησιμοποιούν το, τον ΙΚΑΟ θα ήταν σκοπιμότερο να διατυπώσουν επικοδομητικές προτάσεις για να καταλήξουμε σε μια παγκόσμια συμφωνία η οποία θα θέσει θέσπιζε ίδιους κανόνες, ίσους κανόνες για όλους και θα μας επέτρεπε να έχουμε μια πιο βιώσιμη αερο ναυτιλία. Στη δεύτερη ε, συμφωνία μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών που υπεγράφει τον, που ε, έγινε τον Άνοιξη και αυτή τη στιγμή περνάει από τη διαδικασία της έγκρισης οι Ηνωμένες Πολιτείες στο άρθρο 15 αυτής της συμφωνίας δέχθηκαν ότι τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν και ότι οι επιτροπές πρέπει να δούνε αν εφαρμόζονται διπλά μέτρα και σταθμά και κάποια ε, και ότι πρέπει να αποφευθούν ορισμένα πράγματα. Οι διαπραγματεύσεις προβλέπουν την αμοιβαία αναγνώριση αυτής της εμπορίας εκπομπών. Γι' αυτό απευθύνω ένα σαφές μήνυμα, το οποίο είναι σαφές, σαφέστατο δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Ο κύριος Κράμερ για την ομάδα Παρακαλώ για 1,5 λεπτό. Herr Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για τις αφήσεις σας δηλώσεις. Ελπίζω να μπορέσετε να τις θέσετε και σε εφαρμογή σε, στις διαπραγματεύσεις. Γιατί η Κοπεχάγη ήταν αποτυχία, ήταν καταστροφή γιατί δεν είχε στόχους η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπαιζε το γνωστό παιχνίδι του Μικάντο, όποιος ε, κονηθεί πρώτος ε, χάνει. Αυτή ελπίζω να μην είναι πια η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα ανταλλαγής των εκπομπών ξέρουμε ότι έχει εισαχθεί και έγινε δεκτό από τις αεροπορικέ εταιρείε προκειμένου να αποφευθεί ο φόρος ε, στην κυροζήνη. Ωστόσο 30 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέτουν τα κράτη-μέλη μέσα από τον ε, ε, μέσα από τα, τους προϋπολογισμούς τους μόνο και μόνο, μάλλον χάνουν τους προϋπολογισμούς μόνο και μόνο επειδή υπάρχει αυτή η απώλεια του φόρου της κυροζήνης. Ε, ας αγάγουμε λοιπόν το φόρο κυροζήνης να καταλάβουν ε, πόσα πει διαβάζει ο Σάκος. Μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι εκπομπές καυσαερίων από τα αεροπλάνα και... Ε, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ε, λύσεις, ε, δεν υπάρχουν ποινές εις βάρος των αεροπορικών εταιριών για αποζημίωση του, ε, επιβάτη σε περίπτωση καθυστέρηση. Είναι τρει ώρε το όριο για την αποζημίωση επιβατών, ενώ είναι μία ώρα για τα τρένα. Τι έχουμε δηλαδή παραχαϊδέψει και τελικά δεν θέλουν να εφαρμόσουν ούτε αυτέ τι βασικέ ε, συμφωνίε και αποφάσει. Νομίζω ότι πρέπει αυτό να το, επιβάλλουμε. Τώρα ερχόμαστε στον κατάλογο των εγγεγραμμένων μιλητών. Η κυρία Τσικάο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Η παγκόσμια οικονομία ε, εξαρτάται ε, απόλυτα από τις αεροπορικές μεταφορές. Οι μελέτες που έχουν γίνει έδειξαν ότι το 26% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα οφείλονται στις αεροπορικές μεταφορές. Είναι προφανές πως ε, οι νέες τεχνολογίες θα επιτρέψουν στον περιορισμό αυτών των εκπομπών. Μία πρόσφατη μελέτη που αναφέρεται στην απόδοση των ε, κινητήρων, των αεροσκαφών, δείχνουν μια σημαντική μείωση αυτών των εκπομπών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται συμφωνίες με τρίτες χώρες ε, σχετικά με θέματα των αεροπορικών μεταφορών. Μια τέτοια συμφωνία είναι η συμφωνία που έχει συναυθεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά και τέτοιες συμφωνίες θα πρέπει να περιέχουν διατάξεις οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ε, μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τώρα, ο κανονισμό του 2008 στο άρθρο 25 προβλέπει πως εάν μια τρίτη χώρα υιοθετήσει μέτρα μείωσης ε, των ε, εκπομπών αερίων από πτήσεις που προέρχονται από τη χώρα τους και προσγειώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα φροντίσουμε να ε, ληφθούν και από πλευρά μα ε, τα αντίστοιχα μέτρα. Αυτό το οποίο ζητάμε από την Κομισιόν είναι να μα δώσει κάποια παραδείγματα αυτή τη ελληνεπίδραση ε, που υπάρχει και τα αποτελέσματα αυτών. Τώρα, το άρθρο λοιπόν 25 του 2008 αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουν να καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να κατρύψουν συμφωνία γενικά με την λήψη μέτρων για την μείωση των εκπομπών αερίων. Σύμφωνα με την την ε, με αυτή την συμφωνία δεν ε, θα χρειαστούν να ληφθούν περαιτέρω μετά. Κύριε Επίτροπε, έχει προκληθεί κάποια τροποποίηση. Έχει το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Sorry. <coughs> Hello. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω την υποστήριξή μου σε αυτή την προφορική ερώτηση, γιατί θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο για τις Ηνωμένε Πολιτείε, το Μεξικό και τον Καναδά να προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη συμπερίληψη της αεροπορίας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι από το 2012 αυτό που προβλέπεται να γίνει είναι ανεπαρκές σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να είχαμε εφαρμόσει. Παραδείγματος χάρη, ο τομέας δεν θα, μπορεί να αξιοποιεί ε, μερίδια από άλλους τομείς. Εκ το να συμπεριλάβουμε την αεροπορία είναι εν πάση περιπτώσει ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμπληρώνει ένα νομοθετικό κενό που δεν υπήρχε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αρχή του ρηπαίνων πληρώνει νομίζω ότι ισχύει εδώ περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε και να, τις ε, θέσεις μας και να μην επιτρέψουμε να υπονομεύονται από τρίτες χώρες. Πρέπει η Επιτροπή και το Συμβούλιο να δηλώσουν ότι σκοπεύουν να εφαρμόσουν τον ε, νόμο που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις επικείμενες συνομιλίες. Τώρα ο κύριος θα πάρει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αξιοποιεί την ενέργεια να περιορίσει και να περιορίσει την, σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Είναι αυτό ένα σημαντικό βήμα για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των αεροπορικών πτήσεων και τα μέτρα πρέπει να επεκταθούν και σε τρίτες χώρες των οποίων τα αεροσκάφη πετάνε και προσγειώνονται σε αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι αλλιώς θα υπάρξει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εμείς προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και γι' αυτό πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη στις πράξεις μας. Οι συμφωνίες με τις αεροπορικές εταιρείες τρίτων χωρών Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουν ότι θα ισχύει ο ανταγωνισμό ενώ θα περιορίζονται οι εκπομπέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει συντονιστικά μέτρα και να εξασφαλίσει ότι θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τις τρίτες χώρες. Ε, ο κύριος Κέλλη και ο κύριος Μαρινέσκο έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Κέλλη καταρχάς για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να πω ότι με κατέπληξαν τα όσα άκουσα σήμερα και κατά κάποιο τρόπο με κατέθλιψαν κιόλας. Βλέπω ότι συνεχίζουν τα προβλήματα σχέση με τις εκπομπές των ε, καυσαερίων, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη κρατών όπως ε, η Βραζιλία, η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, που και έχουν υψηλέ εκπομπές αλλά και ακολουθούν τις δικές τους ε, πολιτικέ. με δεδομένο δε τις οικονομικές εξελίξεις, δημογραφικές εξελίξεις, τον αναπτυσσόμενο τουρισμό, την αυξημένη ανάγκη για κινητικότητα, θα πρέπει να διερωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να προσφέρουμε καινοτομία, με, όπως σε παραδείγμα με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τα ε, κτίρια που είναι ενεργειακά σχεδιασμένα. Κάτι αντίστοιχο χρειαζόμαστε και στην αεροπορία. Κύριος Μαρινέσκου. Ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Το να συμπεριληφθεί οι αεροπορικέ μεταφορέ στο σύστημα εμπορία είναι κάτι το θετικό, διότι η νομοθεσία θα πρέπει και αυτή να προσαρμοστεί κατάλληλα. Η οδηγία όσο έχει από το 2012 θα μας διευκολύνει αυτό το έργο. Το αίτημα ε, σε τρίτες χώρες προκειμένου να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αυτό το σύστημα νομίζω ότι δεν είναι κάτι το αποτελεσματικό θα έχει ως αποτέλεσμα να περιορίσει την αγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών και πραγματικά θα πλήξει την προσπάθεια της Ευρώπης στο να καταλήξει σε μια τομεακή συνολική συμφωνία για τη μείωση των ε, της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν το, θα πρέπει η εφαρμογή αυτής της οδηγίας να τύχει εφαρμογή και από τρίτες χώρες. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χάσουμε την, την, τα όσα έχουμε πετύχει στον τομέα και θα διευκολύνουμε την μείωση κατανάλωσης. Ένα λεπτό κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, συμφωνώ ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περιορίσουμε τις εκπομπές όσο γίνεται περισσότερο. Θεσπίζονται τους αναγκαίους κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται και αν οι φίλοι μας από τις Ηνωμένε Πολιτείες δεν θέλουν να το δεχθούν αυτό, εμείς πρέπει να συνεχίζουμε τις επαφές και τις συνομιλίες μαζί τους και έναν διάλογο για να προσπαθώντας να πετύχουμε τους ε, ε, αναγκαίους στόχους. Η ένταξη των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο σύστημα εμπορία δικαιωμάτων δεν θα είναι τόσο μεγάλο βάρο για τη βιομηχανία πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και τα άλλα μεταφορικά μέσα που πρέπει να περιορίσουν και εκείνα τις εκπομπές τους και πρέπει ε, να, να, να ακολουθήσει και το παράδειγμα των άλλων μεταφορικών μέσων και αεροπορία. Τη συζήτηση θα κλείσει ο Επίτροπος, ο κύριος Χάν. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση ε, για τι διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΚΑΟ. μα υποστηρίζει δηλαδή, αν και δεν περιμένω τίποτε διαφορετικό. Σα ευχαριστώ πολύ. Η υποστήριξη που μα προσφέρετε, η υποστήριξη που εκφράστηκε από τη συζήτηση, θα διαβεστεί στην κυρία Χίλγκαρτ και στον Επιτροπό Κάλλα, που έχει το ε, καθήκον να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στη ως προς τις ερωτήσεις που έχουν διατυπωθεί, μπορώ να τις απαντήσω εκ του προχείρου, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά η νομοθεσία, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία έχει εγκριθεί από Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, είναι νομοθεσία την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει προς κάθε ε, παραλείπτη ανεξαρτήτως της υπηκότητας ή της έδρας του. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι και οι, ε, οι εταιρείε από τις ΗΠΑ θα πρέπει να επαχθούν στο σύστημα αυτό. Εάν δεν υπαχθούν θα πρέπει να επιβληθούν απαγορεύσεις πτήσεως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά ως τελική λύση, εφόσον δηλαδή δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις συνθήκες του συστήματος και σε αυτό περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υποστήριξη των κρατών μελών για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων απαγορεύσεις πτήσης. Αυτό το έχουμε και νομικά επαληθεύσει με πολύ μεγάλη προσοχή με βάση και την ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ξέρουμε ότι θα μας ε, δικαιώσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα δεχθεί μία περίπτωση απαλλαγής από το σύστημα των εκπομπών τέτοιου είδους ε, επιχειρήσεων από τρίτα κράτη. Δεν θα δεχθεί δηλαδή τίποτε το οποίο να υπονομεύει το σύστημα ανταλλαγής εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ το πολύ κύριε επίτροπε. έληξε η συζήτηση εδώ.